στις 12. Πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση του κυρίου Ζαντό. Οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών. Εξ του κυρίου Ζαντό, να δώσω το λόγο στην κυρία Φρανσίσκα Κέλλερ. Dear colleagues, it's okay, yes. Now working. Dear colleagues, on behalf of the Συνάδελφοι, εκ μέρου του Δ. Ε, Ζαντό, ο οποίο δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, θα σα μεταφέρω μερικέ σκέψει, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω τη μεγάλη χαρά να ψηφίζουμε αύριο την πρώτη έκθεση τη Κομισιόν για τους Οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων. Η σχετική εργασία ξεκίνησε πριν από πάνω από τρία χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης για την εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτών των τριών τελευταίων χρόνων. Πριν από τρία χρόνια στην Επιτροπή ΙΝΤΑ έφτασε στα χέρια μας ένας φάκελος όσον αφορά τις δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων και το πώς το πλαίσιο λειτουργίας τους θα γίνει νόμος. Μετά από την θέσπιση της συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δοκιμάσει τις δυνάμεις του, συνειδητοποιώντας την ευθύνη του όχι μόνο εναντί των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και εναντί του πνεύματος και του γράμματος της νέας συνθήκης. Ήταν η στιγμή που η οικονομική και χρηματοπιστρική κρίση ξέσπασε στην Ευρώπη και έστρεψε τα φώτα στον τρόπο με τον οποίο ξεδίδουμε τα κονδυλιά μας. Ε, αναρωτήθηκα και εγώ τι γνωρίζουμε για τις δραστηριότητες αυτές των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων που λειτουργούν με χρήματα των φορολογουμένων. Δεν αφισβήτησα τον ρόλο αυτών των οργανισμών, απλώς είπα ότι γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη λειτουργία τους. Επιπλέον, διαπίστωσα ότι οι εθνικοί οργανισμοί και οι απαιτήσει της Λισαβόνας δεν είχαν σχέση μεταξύ τους. Αγνώσαμε δηλαδή την υποχρέωση να υπηρετούν και αυτοί οι οργανισμοί του στόχου τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα τη συνθήκη. Στην Επιτροπή ΙΝΤΑ όλοι συμμερίστηκαν τι θέσει αυτέ, ανεξαρτήτω των διαφωνιών μα. Βρεθήκαμε λοιπόν και σταθήκαμε όλοι ενωμένοι, υπεραμεινόμενοι τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Είχε λοιπόν ομόφωνη υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Και ζήτησαν από την Κομισιόν υποβάλει τη σχετική έκθεση ώστε και οι αναδυόμενες οικονομίες να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την κατάσταση και προσπάθησε να απαντήσει κατά πόσον τα κράτη-μέλη και εθνικοί οργανισμοί συμμορφώνονται με την ανάγκη ακριβώ της πρόθεσης της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Η Κομισιόν έστειλε το μήνυμά μας στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ λοιπόν συναφώς και την Κομισιόν και τον κύριο Ντένις Τεντονές συγκεκριμένα. Η ευρενή ψηφορία αφορά την πρώτη έκθεση της Κομισιόν για τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον αφορά τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή αυτού του εγχειρήματο. Τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται να αποδείξουν πώς αξιοποιούν τα κονδύλια αυτά για την προβολή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή πώς ενσωματώνουν ακριβώ τα θέματα του περιβάλλοντος στις πολιτικές τους. Στην έκθεση λοιπόν γίνονται προτάσεις σχετικά με το πώς θα προωθεί αυτή η προσπάθεια στο μέλλον και πώς η Κομισιόν θα μπορεί να αξιολογεί τις σχετικές εθνικές εκθέσεις. Η επόμενη έκθεση θα είναι σαφώς καλύτερη. Σαφώς ευχαριστώ τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι ένας καλύτερος πρωταγωνιστής παγκοσμίως για τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε μια οικονομική κρίση με την ε, παγκοσμιοποίηση να αυξάνεται συνεχώς, ε, ε, βλέπουμε το ότι καταραίουν διάφοροι μηχανισμοί Γι' αυτό και οι οργανισμοί εξωγικών πιστώσεων ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν, νομίζω, καλύτερα τους, ε, ε τις ε, ανισότητες είτε μεταξύ βορρά και νότου, είτε και τις ε, ανισότητες μεταξύ διαφόρων περιφερειών, περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει βεβαίω σαφής αντίθεση εδώ με τους ε, στόχους που ε, συνεχώς θέλουμε να ε, επιτύχουμε όσοι υπερασπίζονται τον ελεύθερο ανταγωνισμό ό,τι και να συμβεί με κάθε τίμημα χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους ενώ μια αόρατη χείρ μπορεί ξαφνικά να καταστρέψει τον ανταγωνισμό και να καταστρέψει τα πιο αδύναμα συστήματα. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εκ μέρου του Επιτροπού Τεχούχτ, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ δι και δι τον κύριο Ζωτό και τον κύριο Κέλλερ για τι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε απόψει για τι εξαγωγέ πιστώσει. Η παγκόσμια οικονομική κρίση κατέδειξε με τρόπο που δεν έχει προηγούμενο πόσο σημαντική είναι η χρηματοδότηση για τι διεθνεί εμπορικέ ροέ. Οι εξαγωγικέ πιστώσει είναι ζωτική σημασία σε προκειμένου και είναι ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο των προσπαθειών πρόθεσης των ευρωπαϊκών εξαγωγικών συμφερόντων. Η ζωτική σημασία υπάρχει διαφάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το πώς οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων κινούνται. Είναι και ένας από τους στόχους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μεταξύ άλλων και του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων. Αν δούμε την, τον πρωτογύρο υποβολή υποβολής εκθέσεων ε, θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τις απόψεις της τρέχουσας έκθεσης ότι οι εθνικές εκθέσεις παρέσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, αυτές που ζητά ο κανονισμός 1233 του 11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει προσιλωμένη στο άρθρο 21 όσον αφορά την άσκηση των εξωτερικών πολιτικών. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις όσον αφορά τις πολιτικές που αφορούν τις εξαγωγικές πιστώσεις που διατυπώνονται στην έκθεση. Θα λύσουμε περαιτέρω τις θέσεις αυτές και συναρτήσει των συμπερασμάτων θα δούμε πώς θα διατυπωθεί εκ νέου κανονισμός. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη της έκθεσης της Κομισιόν και τις διαρκείς σας προσπάθειες να υποστηρίξουμε τις αναδυόμενες οικονομίες. Καθώς προσπαθούμε να βρίσουμε και μια ομάδα στο θέμα. Η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία στερπίδουν όλο και περισσότερο στο διεθνές εμπόριο. Σχετικώ χρειάζεται διάλογο με τι χώρε αυτέ. Ο Επίτροπος Δεχούχ θα συνεχίσει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι σχετικέ εξελίξει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κλείσαμε λοιπόν και το τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης. Η ψηφοφορία για το το σημείο θα γίνει όπως και οι υπόλοιπε αύριο το πρωί στις 12. Η επόμενη συνεδρίαση ξεκινά αύριο 3η 2 Ιουλίου στις 8.30. Έχει δημοσιευθεί η διάταξη, βρίσκεται